Μετά από ε, το, το ότι η κυρία Μάχ και η κυρία Γκλένις Βίλμοτ παρετήθηκαν, χειρεύουν οι θέσεις τους από την 1η Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου 2017 ε, αντίστοιχα και ενημερώνουμε τις Εθνικές Αρχές. Μετά το διορισμό της κυρίας Μαρία Γκάμπριελ ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κυρίου Χέρμπετ Ρόιλ ως μέλος ε, της ε, Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ρινανίας Άνω και της κυρίας Γκάλ Πέλτς ως μέλος του του δικαστηρίου λαμβάνουμε υπόψη ότι χειρεύουν οι θέσεις τους. Με συγχωρείτε του ελεγκτικού συνεδρίου. Μετά από το διορισμό του κυρίου Λουί Αλιό στο γαλλικό κοινοβούλιο θεωρούμε ότι χειρεύει η θέση του από τις 21 Ιουλίου 2017. η κύριοι ε, Φράνσις Τζάμιτ Ντίμεχ, Ντένις Ράτκε, Τζόναθαν Μπούλοκ και Φρανς ε, Ζαμέ, καθώς και η Βαρόνι Νόσε ε, Μομπάρικ, έχουν διοριστεί και αντικαθιστούν αντιστοίχως τους Κομοντίνη, Κακία Ρόιλ, Χέλμερ, ε, Λουί Αλιό και Ντάνκαν. Καλωσορίζουμε τους συναδέλφους και φυσικά τους ΔΙΕΠ